Ladies and once more, please be seated. Καθίστε, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην απογευματινή μας ε, συνεδρίαση. Είναι το τελευταίο ουσιαστικό σημείο της ημερήσιας διάταξης. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα, μας απασχολεί συνεχώς, δηλαδή η κατάσταση ασφαλείας στο Ιράκ και είναι χαρά μου που καλωσορίζω εδώ τα μέλη του πάνελ. Πρώτα απ' όλα η κυρία Ρόζα Μαρία Τζίλη, η οποία είναι υπό διευθύντρια στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, για τις χώρες ε, του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, το Ιράκ και την Ιεμένη. Και μετά είναι ο κύριος ε, Καβα Χασάν, διευθυντής για την Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική στο Ινστιτούτο East West. Κυρίες και κύριοι, το Ιράκ ε, είναι σημαντικό θέμα. Με απόφαση των συντονιστών η Επιτροπή μας θα ταξιδέψει στη χώρα εντός του έτους. Είναι νομίζω επίκαιρο λοιπόν. Και θα ήθελα τώρα να δώσω τον λόγο στην κυρία Τζίλη και μετά στον κύριο Χασάν. Κυρία Τζίλη, έχετε τον λόγο. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Μου είπαν ότι κάποιοι από εσάς θα πάτε στη χώρα φέτος. Νομίζω πως ε, το πιο χρήσιμο θα ήταν να σας αναφέρω κάποια σημεία της ανάλυσής μας για τις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ιράκ αυτή τη στιγμή. Και βεβαίως ε, δεν θα σας προξενήσει η ότι τελικά μάλλον θα δημιουργηθούν περισσότερα ερωτήματα από όσα θα απαντήσω, αλλά ο στόχος είναι να βρείτε μόνοι σας τις απαντήσεις όταν θα πάτε στη χώρα. θα οργανώσω το σκεπτικό μου γύρω από δύο πράγματα. Είναι, υπάρχουν οι προφανείς προκλήσεις ασφαλείας αυτή τη στιγμή στη χώρα, το ΝΤΑΕΣ, το Ισλαμικό κράτος, αλλά και πιο μακροπρόθεσμες προκλήσεις. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι Το ΝΤΑΕΣ, σύμφωνα με την ανάλυση μας, είναι ένα σύμπτωμα το οποίο βεβαίως ε, μπόρεσε να αναπτυχθεί λόγω της πραγματικότητας που υπάρχει στη χώρα. Και μετά θα αναφερθώ σε αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε τις αιτίες που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα και μέσω μικρό πρόθεσμα. Θα ξεκινήσω με μια θετική ανάλυση όσον αφορά τη μάχη κατά του ΝΤΑΕΣ. Υπάρχει μια γενική αισιοδοξία όσον αφορά τη στρατιωτική πρόοδο. Τα γεγονότα είναι ξεκάθαρα. 40% της επικράτειας που ήταν στα χέρια του ΝΤΑΕΣ το 2014 έχει απελευθερωθεί. Έχουμε κάποιες ε, πρόσφατες ε, σημαντικές εξελίξεις με την απελευθέρωση της Ραμάντη και της Φαλούτζας και της ε, Καϊάρα που είναι 60 χιλιόμετρα από την Μουσούλη κάτι το οποίο αυξάνει τις εικασίες ότι η Μοσούλη θα μπορούσε ίσως να αποτελέσει αντικείμενο εκστρατεία φέτος, στόχο εκστρατεία. Και βεβαίως βλέπουμε ότι υπάρχει ακόμα ρόλος της συμμαχίας που συμβουλεύει και εκπαιδεύει τα Ιρακινά στρατεύματα. Έχουμε λοιπόν σαφώς πρόοδο που αναγνωρίζεται γενικώς και μπορούμε να είμαστε αρκετά αισιόδοξοι ότι αυτή τη στιγμή το αν θα νικηθεί το ΤΑΕΣ είναι ζήτημα χρόνου και όχι ένα πραγματικό ερώτημα. Βεβαίως η Μοσούλη είναι το επόμενο μεγάλο βήμα. Η Μοσούλη είναι νομίζω μια καλή αφορμή για να περάσουμε στις ε, μακροπρόθεσμες ε, προκλήσεις ασφαλείας της χώρας. Γιατί η απελευθέρωση της Μοσούλης θα είναι και μια μεγάλη ευκαιρία και είναι συμβολική η πόλη αλλά είναι και τεράστια πρόκληση πολλά από τα όσα θα συμβούν στη χώρα μακροπρόθεσμα συνδέονται με το πώς θα εξελιχθεί η απελευθέρωση της Μοσούλης. Όταν μιλάμε για απελευθέρωση περιοχών, κατευθείαν περνάμε στις μακροπρόθεσμες ε, προκλήσεις. Όπως είπα, το είναι ένα σήμα, αν θέλετε, εμπορικό, το οποίο ε, πέτυχε λόγω της ε, κατάστασης στην χώρα. Η μεγάλη πρόκληση λοιπόν είναι η σταθεροποίηση της χώρας. Μιλάμε για τις απελευθερωμένες περιοχές και εκεί πέρα ακριβώς θα δούμε όλες αυτές τις μεσομακροπρόθεσμες ε, προκλήσεις. Κάθε περιοχή είναι διαφορετική έχουμε τους ε, απελευθερωμένους λαούς ε, και περιοχές και τους απελευθερωτές ε, και ακριβώς το πώς θα τα πάνε όλοι αυτοί μεταξύ τους είναι η μεγαλύτερη πρόκληση ασφαλείας για την χώρα και υπάρχει κάτι το οποίο είναι εκπληκτικό και εμένα προσωπικά με εξέπληξε όταν πήγα τον Αύγουστο του 2014 στην χώρα ότι ενώ θα μπορούσαμε να περιμένουμε ότι ο κοινό εχθρός και η κοινή πρόκληση θα ένωνε τη χώρα, αυτό το οποίο είδαμε είναι μια χώρα όπου υπάρχουν ε, έθνο-θρησκευτικές ε, συγκρούσεις και μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων αλλά και εντός των διαφόρων κοινοτήτων. Και η πολιτική κρίση την οποία ζούμε τους τελευταίους μήνες είναι απλά αποτέλεσμα αυτού. Αυτή τη στιγμή η χώρα χρειάζεται πολιτική σταθερότητα για να κάνει αυτές τις ε, μεταρρυθμίσεις που θα αντιμετωπίσουν τις αιτίε που προκάλεσαν την άνοδο ακραίων ομάδων και μόνο έτσι θα υπάρξει μακροπρόθεσμη σταθεροποίηση. Επίσης, όταν μιλάμε για τις απελευθερωμένες περιοχές ε, και λαούς, πρέπει βεβαίως να δούμε και την δυσαρέσκεια των διαφόρων μειονοτήτων και της μεγαλύτερης μειονότητας ε, των Σουνιτών που είναι ένας λόγος ε, για τον οποίο ήταν ε, επιτυχές το ΝΤΑΕΣ. Είναι περίπλοκα τα ζητήματα, όλοι θυμόμαστε το 2014 τα ερωτήματα για τον ρόλο των ντόπιων και την επιφυλακτικότητα που υπήρχε μεταξύ του πληθυσμού. Αλλά ανέφερε και τους απελευθερωτές. Και εδώ φτάνουμε σε μια άλλη θεμελιώδη πρόκληση ασφαλείας, το ότι δηλαδή η χώρα είναι πολύ στρατιωτικοποιημένη. Έχουμε το PMF, τους Πεσμεργά, διάφορες ε, φιλετικές ε, πολιτοφυλακές, διάφορες δυνάμεις που έπρεπε να ε, χρησιμοποιηθούν, να αναδιοργανηθούν και να χρησιμοποιηθούν λόγω του κοινού εχθρού του Και το πώς τώρα θα ενταχθούν όλοι αυτοί σε έναν εθνικό στρατό η μεταρρύθμιση αυτή του τομέα της ασφαλείας είναι πολύ βασικό ζήτημα για την σταθεροποίηση της χώρας και για την μακροπρόθεσμη σταθερότητα. Θα τελειώσω λέγοντας το τι προσπαθεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια κατάσταση που είναι πολύ περίπλοκη. Είμαστε πεπισμένοι ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τη μόνη δυνατή επιλογή, δηλαδή να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε την τωρινή κυβέρνηση σε μια επιχείρηση οικοδόμησης κράτους. Θεωρούμε πως η ενότητα και η εδαφική ακεραιότητα είναι η μόνη επιλογή για τη χώρα και καλούμε και την κεντρική διοίκηση και τις περιφερειακές διοικήσεις να συνεργαστούν ακόμη περισσότερο και να οικοδομήσουν μαζί μια ισχυρή χώρα. Λοιπόν, συμφωνούμε όλοι ότι χρειαζόμαστε ένα ισχυρό κεντρικό κράτος αλλά πρέπει μετά να υπάρξει ένας μηχανισμός αυτονομίας και αποκέντρωσης, γιατί βλέπουμε ότι το μέλλον της χώρας δεν έχει άλλη επιλογή ουσιαστικά. Επίσης θεωρούμε πως ένα άλλο σοβαρό κομμάτι των μεταρρυθμίσεων είναι οι μεταρρυθμίσεις όπως είπα στον τομέα της ασφάλειας που δεν είναι εύκολες και είναι ακόμη πιο δύσκολες στην κατάσταση όπως έχει τώρα, αλλά είναι σαφώς η μεταρρύθμιση αυτή που έχει σημασία για τη σταθεροποίηση της χώρας. Προσπαθούμε λοιπόν να στηρίξουμε την κυβέρνηση που υπάρχει και οπωσδήποτε μας ενθαρρύνει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που προτάθηκε από την κυβέρνηση το 2014. Γνωρίζουμε ότι τα πράγματα δεν πάνε ε, τόσο καλά από πολιτική σκοπιά όσο από στρατιωτική, αλλά επιμένουμε ότι η στρατιωτική λύση δεν θα είναι μακροπρόθεσμη λύση. Οπότε θέλουμε να γίνουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις και να υπάρξει ένας πραγματικός μηχανισμός συμφιλίωσης για τη χώρα. Και βεβαίως μια που πρέπει να σκεφτούμε μέσω μακροπρόθεσμα αλλά έχουμε βεβαίως και τα άμεσα μπροστά μας προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό αντιμετώπισης της κατάστασης. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3,5 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένοι και περιορισμένοι πόροι και βεβαίως δεν ξέρουμε τι θα γίνει από την ε, πιθανή μάχη της Μοσούλης. Οπωσδήποτε και στο δεύτερο γύρο θα μας πείτε κι άλλα. Τώρα ο κύριος Χασάν έχει το λόγο. Thank you very much. Ε, Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την πρόσκληση. Κυρίε και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Με την απελευθέρωση της Φαλούτζα και με την επανακατάληψη της Αλφαγιάρα ο πόλεμος κατά του ISIS μπαίνει σε μια κρίσιμη φάση. Σύμφωνα με το HIS από τις 4 Ιουλίου φέτος ε, ο ISIS ελέγχει γύρω στις 6.300 τετραγωνικά χιλιόμετρα περίπου, δηλαδή όσο η Δυτική Βιργίνια, η Δυτική Virginia ή η Ιρλανδία. Έχασε 40% των εδαφών του το ISIS και στους τελευταίους 6 μήνες υπήρξε μια περαιτέρω μείωση τάξεις 12%. Ε, αδιαφεσβήτητα όλα αυτά είναι καλά νέα και πρέπει ε, να τα ε, δεχτούμε ως τέτοια. Όμως καθώς προετοιμαζόμαστε για την κρίσιμη μάχη της Μοσούλης ε, είναι μεγάλες προκλήσεις για την συμμαχία κατά του ISIS. Πρώτα απ' όλα, παρότι η συνάντησή μας αφορά τα ζητήματα ασφάλειας στο Ιράκ, κατά τη γνώμη μου είναι απαραίτητο να μην ξεχνάμε ε, τη μάχη των ιδεών μεταξύ του ISIS και του υπόλοιπου κόσμου. Η φρικτή τελευταία ε, επίθεση στην Βαγδάτη αλλά και στην Μπαγκλαντές, στην Τάκα, στην Κωνσταντινούπολη ε, μας υπενθυμίζουν κατά τρομερό τρόπο την επιμονή αυτής της ιδεολογίας, την, την ανθεκτικότητα αυτής της ιδεολογίας του ISIS. Ο ISIS λοιπόν χάνει, χάνει έδαφος αλλά κερδίζει σε ιδέες, τουλάχιστον για την ώρα μετά την στρατιωτική ήττα του ISIS θα πρέπει να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια εναλλακτική αφήγηση για τους ε, στρατιώτες του ISIS που έρχονται από περίπου 100 χώρες ε, μεταξύ των οποίων και το Βέλγιο η έλξη που υπάρχει ε, προς τον ISIS δεν είναι θέμα του Ιράκ είναι παγκόσμιο πρόβλημα η παγκοσμιοποίηση του ISIS πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω της παγκοσμιοποίησης της αλληλεγγύης όλα τα θύματα της βαρβαρότητας του ISIS ε, πρέπει να δεχθούν την αλληλεγγύη αυτή. Ένα από τα πιο ισχυρά μηνύματα στα κοινωνικά μέσα ε, στο Ιράκ είχε να κάνει με την έλλειψη ε, δειγμάτων αλληλεγγύης ανά τον κόσμο μετά την ε, τρομερή επίθεση στη Βαγδάτη, σε, αν το συγκρίνει κανείς με τις επιθέσεις της Βρυξέλλης στο Παρίσι. Δεύτερον, κατά την απελευθέρωση της Φαλούτζα υπήρξαν παραβιώσεις των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Σύμφωνα με τη Human Rights Watch, αλλά και έρευνες της κυβέρνησης του Ιράκ, υπήρξαν ε, ε, παραβιάσεις δικαιωμάτων που κρύβονται. Πρέπει να γίνουν λοιπόν οι έρευνες και πρέπει όσοι έχουν παραβιάσει τα ανθρώπινα δικαιώματα να λογοδοτήσουν προς τα θύματα και τις οικογένειές τους. Παρότι βεβαίως ο Άισις είναι αυτός που έκανε την επίθεση στο, στην αγορά της Καράντα, ε, σχετίζεται και με τον καταγραμματισμό και τη διέρεση που υπάρχει στις αστυνομικές και στρατιωτικέ δυνάμεις του Ιράκ. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Ελέγχθηκε προηγουμένω. Στη Βαγδάτη αυτέ οι δυνάμει, οι δυνάμει του Ιράκ δηλαδή, είναι χωρισμένε μεταξύ του Ιρακινού στρατού, του Υπουργείου Ιστορικών, δύο υπηρεσιών πληροφοριών, ε, δυνάμει ε, κοινωνική, ε, λαϊκές, μάλλον, ε, λαϊκής πολιτοφυλακής, καθώς και περιπολίες γειτονιάς όλες αυτές οι δυνάμεις έχουν τον ίδιο στόχο. Να, να υπερασπιστούν τη Βαγδάτη. Να υπερασπίσουν τη Βαγδάτη. Ο πολλαπλασιασμός των διαφόρων υπηρεσιών, η επικάλυψη ευθυνών δημιουργεί σύγχυση, δημιουργεί χάος, δημιουργεί έλλειψη συντονισμού. Το αποτέλεσμα είναι ότι ορισμένε φορές είναι δύσκολο να λογοδοτήσουν οι κάποιες υπηρεσίες όταν γίνουν τρομοκρατικές επιθέσεις όπως τώρα. Η κατάσταση είναι καλύτερη στο Ιρακινό Κουρδιστάν ε, σε σχέση με το υπόλοιπο Ιράκ, αλλά και εκεί υπάρχουν ζητήματα ασφάλεια. Παρά τις υποσχέσεις για μεταρρυθμίσεις και παρά τα σχέδια των Κούρδων ε, ηγετών να μετατρέψουν τις υπηρεσίε ασφαλείας και του πεσμεργά σε θεσμικές ε, δυνάμεις, εξακολουθούν να χωρίζονται κομματικά μεταξύ KPD και PUK. Το Κυρκούρκ αλλά και άλλα αμφιλεγόμενα εδάφη ε, στο, στα βόρεια της Βαγδάτης ε, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό των πολλών και διάφορων ε, δυνάμεων ασφάλειας. Εκεί όπου είχαμε τη γενοκτονία κατά τον Γιαζίντη, το PKK και το PUD έχουν ξεκινήσει μια σύραξη η οποία είναι καταστροφική για όλους. Αυτή η εσωτερική διαμάχη μεταξύ KBD και PKK και PKK έχει ε, μπλοκάρει τους Γιαζίντι και την επιστροφή τους ε, στην χώρα τους. Δεν περίμεναν αυτό οι Γιαζίντι όταν ε, είχαν αποφασίσει να επιστρέψουν στον τόπο τους. Αυτές οι διαθροτικές δομές δεν προϊονίζουν τίποτα θετικό σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του ISIS και ιδιαίτερα την απελευθέρωση της Μοσούλης. Υπάρχουν υπαξιακά ζητήματα στο τι θα γίνει μετά και πρέπει να αντιμετωπιστούν τώρα και όχι αργότερα. Ποιο θα ελέγξει ποιο μέρο τη πόλη, ποιε δυνάμει μπορούν να γίνουν αποδεκτέ βεβαίω από τι τοπικέ κοινωνίε και να παράσχουν ασφάλεια, ποιοι θα συνεισφέρουν στην ανοικοδόμηση και ποιοι θα του ελέγξουν. Ποιο θα είναι το μέλλον των αμφιλεγόμενων ε, ε εδαφών διαμάχης μεταξύ Σουνιτών και Κούρδων. Ε, επίσης υπάρχει ένας πολιτικός καταγερματισμός που αποτυπώνεται επί τόπου. Οι μεγάλες ε, Ιρακινές κοινότητες και τα κόμματα είναι ε, διαιρεμένα σε αφορά το μέλλον του Ιρακινού κράτους. Το πολιτικό σύστημα που προέκυψε μετά το 2003, μετά την κατάρρευση του Σαντάμ Χουσέιν, καταραίει τώρα μπροστά στα μάτια μας. Οι κοινότητες είναι χωρισμένες και στο εσωτερικό τους και εξωτερικά. Εσωτερικά δεν υπάρχει συνένεση σε ό,τι αφορά το τι είδους κράτους θέλουν για το Ιράκ μετά το ISIS. Στο εξωτερικό δεν υπάρχει συνένεση σε ό,τι αφορά τη μορφή που θα πάρει αυτό το κράτος με τις άλλες κοινότητες. Οι τελευταίες διαμαρτυρίες, ε, διαδηλώσεις ε, στη Βαγδάτη και η επίθεση στο Κοινοβούλιο χωρίς προηγούμενο δείχνουν ότι υπάρχει ανάγκη μεταρρύθμισης και ότι υπάρχει πολύ σημαντική πολιτική ανταπαράθεση μεταξύ των Σιητών για το τι θα γίνει με το Ιρακινό κράτος μετά το ISIS. Και οι Σουνίτες είναι διαιρεμένοι για το ζήτημα αυτό. Η πολιτική διαδικασία στο Κουρδιστάν ε, έχει φτάσει σε εμπλοκή πολλαπλώς. Το Κοινοβούλιο έχει παραλύσει, δεν μπορούν να συμφωνήσουν τα κόμματα για το μέλλον της περιοχής, για τον Ομοσπονδιακό Ιράκ. Επιπλέον, οι Κούρδοι δεν μπορούν να συμφωνήσουν για ένα μεταβατικό σχέδιο έως τις επόμενες εκλογές που θα γίνουν το 2017. Διότι λίγη η Προεδρία του Μπετζάνη Και βεβαίως τη μεταρρύθμιση του πολιτικού συστήματος. Ούτε εκεί υπάρχει συμφωνία. Κατά πόσο πρέπει να είναι κοινοβουλευτική, ε, προεδρική ή, ή μη προεδρική ε, η, η δημοκρατία. Οι μεταρρυθμίσει, η αντιμετώπιση τη διαφθοράς δεν προχωρούν. Δεν έχει γίνει κάτι σοβαρό προς την κατεύθυνση αυτή, δυστυχώς. Ε, επίσης, επειδή μειώνονται οι τιμές του πετρελαίου, η διαρθρωτική ε, διαφθορά, ε, ο νεποτισμός ε, συνεχίζονται. Το Ιράκ αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση από το 2003 και μετά. Η οικονομική ύφεση επηρεάζει και τον πόλεμο κρατού ISIS. Χρειάζεται λοιπόν το Ιράκ σημαντική οικονομική ενίσχυση, διεθνή ενίσχυση, έτσι ώστε να μπορέσουν να επανέλθουν οι, τα εκατομμύρια εκτοπισμένων στον τόπο τους και να, ξεκινήσουν, να, ξεκινήσει η ανοικοδόμηση. Μπορεί ο ISIS λοιπόν να είναι πολύ κοντά στην οριστική στρατιωτική ήττα, Εάν δεν επιληθούν όμως τα οικονομικά, πολιτικά και στρατιωτικά ζητήματα, δεν θα προχωρήσουμε είναι σημαντικό οι ηγέτες του Ιράκ να πάρουν τα ίνια σε αυτή την προσπάθεια και να δημιουργηθεί ένα νέο πολιτικό σύμφωνο, μια νέα πολιτική συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί εδώ να παίξει ρόλο στη διαδικασία αυτή και πρέπει να παίξει ρόλο. Να βοηθήσουμε τους Ιρακινούς να ε, νικήσουν τον ISIS, να δημιουργήσουν ένα νέο Ιράκ. Πρέπει το Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τις ΗΠΑ, τα Ηνωμένα Έθνη να παίξουν ρόλο δημοσιολαβητή μεταξύ των διαφόρων Ιρακινών ε, πλευρών να πάρουν τι απαραίτητε οικονομικές ε, πρωτοβουλίε έτσι ώστε να βρεθούν κοινά σημεία μεταξύ των Ιρακινών ηγετών. Χρειάζονται αμοιβαίοι συμβιβασμοί. Αυτή η υποστήριξη όμως πρέπει να δίνεται υπό όρους. Πρέπει να βασίζεται σε βασικές δημοκρατικές αρχές. Πραγματικό μοίρασμα των εξουσιών, πραγματικές μεταρρυθμίσεις, κράτος δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα, αντιμετώπιση της παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαφάνεια, λογοδοσία. Χωρίς ε, αυτά τα στοιχεία το νέο Ιράκ θα είναι ίδιο με το παλαιό Ιράκ και ο Άισις θα επιστρέψει πιο βίαιο και πιο εκδικητικό. Πιο βίαιος και πιο εκδικητικός. Σας ευχαριστώ και περιμένω τα ερωτήματά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις δύο πολύ ενδιαφέρουσες ε, παρουσιάσεις και μπορούμε να ξεκινήσουμε έτσι και τη συζήτησή μας. Δεν έχω σημειώσει ακόμα τα ονόματα όσων θέλουν να πάρουν το λόγο. Ας μας το πείτε αν θέλετε να πάρετε το λόγο, να θέσω εγώ πρώτη κάποια ερωτήματα. Σίγουρα αυτά τα οποία ακούσαμε είναι πολύ θετικά. Σε σχέση δηλαδή με την απελευθέρωση πάρα πολλών εδαφών από τον άμεσο έλεγχο του Ισλαμικού κράτους. Σίγουρα όμως δεν μπορούμε να αφήσουμε κανένα γεωγραφικό κενό αυτή τη στιγμή, διότι αν επιτρέψουμε οποιοδήποτε κενό εξουσία το ISIS θα επιστρέψει στις περιοχές αυτές. Αυτό καταλαβαίνουμε και όλες από την ανάλυση που κάνατε και οι δυο σας. Επίσης πραγματικά χρησιμοποιούμε όλες τις δυνατότητες χρηματοδότησης προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε επιτόπου επιχειρήσεις και έχουμε ασχοληθεί καθόλου με τη δυνατότητα να ανακόψουμε τη χρηματοδότηση της ίδιας της ISIS προκειμένου να μην χρησιμοποιήσουν υφιστάμενους πόρους για να πάνε σε άλλες περιοχές, για παράδειγμα στην Συρία, να κινηθούν προς τη Λιβύη. Και μια ακόμα ερώτηση, απευθύνομαι και στους δυο σας πώς αναλύεται την ικανότητα της Ιρακινής κυβέρνησης να έχει μία πολιτική η οποία να μην περιλαμβάνει αποκλισμούς διαφόρων εθνοτικών ομάδων. Το είχαμε πει αυτό και σε μια συζήτηση που είχαμε κάνει ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από λίγο καιρό, ότι θέλαμε δηλαδή πολιτικές ενσωμάτωσης ένταξης όπου να μην υπάρχουν ε, αποκλεισμοί συγκεκριμένων μονάδων. Προφανώς έχουμε δει πάρα πολλές ε, βαρβαρότητες και φρικαλαιότητες στο Ιράκ στα πλαίσια της Υποπιτροπής ε, Άμυνας και Ασφάλειας πολύ συχνά κάνουμε δηλώσεις μετά από τρομοκρατικές επιθέσεις και προσπαθούμε να μην αναφερόμαστε μόνο βέβαια στις τρομοκρατικές επιθέσεις που λαμβάνουν χώρα στην ευρωπαϊκή επικράτεια, αλλά προσπαθούμε να αναφερόμαστε και να αναλύουμε τις απειλές και σε άλλες περιοχές του κόσμου και συγκεκριμένα βέβαια στο Ιράκ. Και μας έχουν απασχολήσει και οι πρόσφατες αυτές επιθέσεις. Από τη μία πλευρά βλέπουμε ότι έχουμε επιτυχίες στις μάχες που διεξάγουμε. Από την άλλη όμως μέσω των τρομοκρατικών αυτών επιθέσεων βλέπουμε ότι ε, η ISIS μπορεί να ανακάμψει και ότι είναι σε θέση να εκδικείται. Μήπως να ξεκινούσαμε με τις ερωτήσεις αυτές και είμαι σίγουρο ότι θα ακούσουμε και άλλες ερωτήσεις από τους συναδέλφους. Ή ας ακούσουμε μάλλον πρώτα κάποιες άλλες ερωτήσεις και μετά θα απαντήσει το κύριο Σέλερ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία ερώτηση που απευθύνω και στους δύο μιλητές ως προς την ανάγκη να δούμε στην πράξη τι μπορεί να γίνει με αυτό το κατακαιρματισμό που είπατε όσον αφορά τις στρατιωτικές δυνάμεις που καταπολεμούν το Ισλαμικό κράτος. Στην πράξη μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μία κατάρρευση του στρατού του Ιράκ. Και από στρατηγικής πλευράς ποια είναι η επιρροή από το Ιράν. Δεν θα έλεγα ότι φταίνε τόσο πολύ οι διάφορες παραστρατιωτικές δυνάμεις, αλλά περισσότερο η διοίκηση από τη συντική περισσότερο πλευρά. Μήπως θα μπορούσαμε να είχαμε μια πιο θετική επίδραση από την πλευρά του Ιράν. Να δούμε δηλαδή πώς θα μπορούσε το Ιράν και οι εκεί στρατιωτικές δυνάμεις να επηρεάσουν την κατάσταση. Γιατί νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε πλέον για κοινή στρατιωτική διοίκηση, αλλά περισσότερο για έναν κατακαιρματισμό. Θέλουμε λοιπόν να γνωρίσουμε περισσότερο ποια μπορεί να είναι επιρροή από την πλευρά του Ιράν. Ισχύει κάτι τέτοιο. Και μπορούμε να πούμε για παράδειγμα ότι μέσα στο επόμενο έτος οι παροστηθικές οργανώσεις θα αρχίσουν να υποχωρούν και ότι θα επικρατήσει περισσότερο επίσημος στρατός του Ιράκ. Και σίγουρα βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι έχουμε έντονα φαινόμενα ρίζοσπαστικοποίησης και βλέπουμε και πάρα πολλές τρομοκρατικές πράξεις ε, του Ισλαμικού κράτους. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι είχαμε τα πρώτα χρόνια συγκεκριμένους αξιωματικούς του Σαντάμ Χουσέιν που χάσαν πια τη δουλειά τους ε, και που ε, πολλές φορές αυτοί συνέβαλαν τελικά στις πρώτες σημαντικές επιτυχίες του Ισλαμικού κράτους. Αναφέρομαι ουσιαστικά σε Σουνίτες αξιωματικούς. Αν λοιπόν έχουμε στρατιωτική ήττα του Ισλαμικού κράτους, ωραία, από πρακτικής πλευράς θα πληγεί πολύ το Ισλαμικό κράτος, αλλά τι γίνεται από ιδεολογικής πλευράς. και ποια εναλλακτική θα έχουμε απέναντι στο ότι στα πλαίσια του Ισλαμικού κράτους υπάρχει μια ισχυρή ραχοκοκαλιά η οποία παρτίζεται ακόμα από Σουνίτες αξιωματικούς. Τι θα απογίνει λοιπόν ακόμα και αν ιτηθεί το Ισλαμικό κράτος, εφόσον τα στοιχεία αυτά θα παραμείνουν στο Ιράκ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε να ευχαριστήσω τους δύο μιλητές μας για όλες αυτές τις πολύτιμες πληροφορίες που μας δώσανε. Τα όσα μας είπατε καταδεικνύουν ότι η μάχη κατά του Ισλαμικού κράτους σημειώνει μια κάποια πρόοδο. Έχω να κάνω κάποιες ερωτήσεις γενικής φύσης και θα ήθελα να μου δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες για κάποιους τομείς που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικοί, με ενδιαφέρον ιδιαίτερα να συνεχίσω εκεί πέρα που σταμάτησε ο προλή σας. θέτει το ζήτημα της ικανότητας του Ισλαμικού στρατού, συγγνώμη, του Ιρακινού στρατού να αναλάβει δράση. Εδώ και 12 χρόνια ρίχνουμε χρήματα στον στρατό αυτό, στον στρατό του Ιράκ, ευρωπαϊκά κονδύλια που έχουν πάει στην κατάρτιση του στρατού αυτού, στον εξοπλισμό αφού του στρατού και το καθεξής. Τα γνωρίζετε όλα αυτά. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το ακόλουθο. Έχουμε τα αποτελέσματα. Εγώ εργαζόμουν στον στρατό της Πολωνίας στο παρελθόν και είχαμε αναλάβει τότε και την κατάρτιση ενός τμήματος του Ιρακινού στρατού και είχαμε αναλάβει την εκπαίδευση μέχρι και 10.000 στρατιωτών σε μια φάση. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί λαμβάνουν από εμά μια κατάρτιση, όλα μπαίνουν αισίω, αλλά στη συνέχεια δεν γνωρίζουμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Θεωρητικά βλέπουμε ότι χιλιάδες άνθρωποι εκπαιδεύτηκαν στα πλαίσια του Ιρακινού στρατού και στη συνέχεια βλέπουμε ότι δεν είναι σε θέση να προστατεύσουν την ίδια τη χώρα τους. Ποια είναι λοιπόν η πραγματική ποιότητα, αν θέλετε, αυτού του στρατού, γιατί εμεί δαπανούμε πάρα πολλού ευρωπαϊκού πόρου, επενδύουμε στην κατάρτιση αυτού του στρατού και δεν βλέπουμε αυτά αποτελέσματα όμω στο τέλο. Και πολύ συχνά βλέπουμε μάλιστα ότι φεύγουν από τον Ιρακινό στρατό και πηγαίνουν με τον εχθρό. Τι κάνουμε λοιπόν. Έχουμε αξιολογήσει καθόλου την τις ποιοτικέ στρατιωτικές ικανότητες του Ιρακινού στρατού. Και μία ακόμα ερώτηση, το βόρειο της χώρας, το βόρειο τμήμα της χώρας, αναφέρομαι στη Μοσούλη και σε άλλες περιοχές, όπου στο παρελθόν υπήρχε μια κάποια σταθερότητα. Οι Κούρδοι εκεί κατάφερναν να διευθετήσουν κάπως τα πράγματα, αλλά σήμερα βλέπουμε ότι ακόμα και αυτή η περιοχή έχει γίνει ο χειρό τελικά της Άισης. Πώς αξιολογείται λοιπόν εσείς την κατάσταση στο βόρειο τμήμα της χώρας. Είναι σε θέση αυτή τη στιγμή οι Κούρδοι να δημιουργήσουν εκεί ένα καθεστώς αυτονομίας, δέχονται υποστήριξη από κάποιους άλλους. Μπορούμε με τον έναν τον άλλο τρόπο να εγγυηθούμε τη σταθερότητα, αν μη τι άλλο, αυτού του τμήματος της χώρας το οποίο είναι κρίσιμη σημασία, γιατί εκεί πέρα έχουμε τα περισσότερα κοιτάσματα πετρελαίου. Οπότε είναι ένα τμήμα τη χώρα που συμβάλλει πάρα πολύ στην οικονομική ανάπτυξη και σταθερότητα τη χώρα. Ευχαριστώ κύριε Φρόντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι προφανές σε όσους παρακολουθούμε τι ειδήσει ε, από το Ιράκ σε τακτική βάση ότι η χώρα είναι σε μαύρο χάλι πολιτικά μιλώντας. Ε, ακόμη χειρότερη κατάσταση για τον πληθυσμό. Γιατί δεν έχει τα βασικά ενός ε, κράτους ε, που λειτουργεί. Από την άλλη, παρενθετικά θα ήθελα να προσθέσω ότι δεν ξέρουμε ακριβώς πώς τα πάει η χώρα, γιατί μόνο τις άσχημες ειδήσει μαθαίνουμε. Υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις σε πολλές ε, χώρες. Ε, όταν είχα πάει στην Ουάσιγκτον, μου λέγανε φίλοι μου, μα θα πας στην Ουάσιγκτον, δεν φοβάσαι μη σε σφάξουνε, ε, έχει τόσους φόνους. Α, δηλαδή αυτό ήξεραν για την Ουάσιγκτον. Αυτό και ότι είναι η πρωτεύουσα, εντάξει. Αυτά έτσι είναι η δισαγωγή αν θέλετε, αλλά το ερώτημά μου αφορά την έκθεση Τσίλκοτ που βγήκε τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου η... διαβάσαμε ότι η κυβέρνηση Τόνι Μπλερ συνεργάστηκε με τις ΗΠΑ για τον πόλεμο του Ιράκ το 2003 και αυτό το οποίο με εξέπληξε ήταν πως ο Τόνι Μπλερ υπερασπίστηκε αυτόν λέγοντας περίπου ότι το Ιράκ είναι καλύτερα τώρα από ότι ήταν επί Χουσέιν. Και χωρίς να ασκήσω κριτική, θα ήθελα να μου πείτε εσείς που έχετε σοβαρή και περισσότερη γνώση από μένα. Ισχύει αυτή η αξιολόγηση αν και δεν ξέρουμε βεβαίως ε, τι θα γινόταν τα τελευταία 13 χρόνια εάν κυβερνούσε ο Σαντάμ Χουσίν. Απλά θα ήθελα να κάνετε μια σύγκριση για τη ζωή των ανθρώπων τότε και τώρα. Σας ε, ευχαριστώ, κύριε Σνάρτ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το Ιράν είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την μάχη κατά του Ισλαμικού κράτους στο Ιράκ. Εγώ συνόδευσα τις δυνάμεις του Σέιμπ από, από τη Βαγδάτη στο Μπέιζι και δεν υπήρχε ούτε ένα στρατιώτης του Ιρακινού στρατού. Όλοι όσοι ανέκτησαν τα εδάφη ήταν, ήταν από τη Χεσμολάχ ήταν από τις ε, τι τις λαϊκές. Στην πραγματικότητα λοιπόν, όχι στην... για ένα πραγματικό ερακινό κράτος, με ένα στρατό, χωρίς πολιτοφυλακές, διότι οποιαδήποτε πολιτοφυλακή είναι ε, εξορισμού ε, αρνητική για ένα κράτος. Οι δυνάμεις ε, του στρατηγού Σουλεϊμάν και δυνάμει Αλκούτς που αποτελούν ε, τις δυνάμεις αντίστασης στο Ισλαμικό Κράτο είναι παράγοντα σταθεροποίηση και χωρί αυτού θα ήταν ήδη στη Βαγδάτη το Άισι. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Μιλάμε για του Κούρδου ω μια, μια σημαντική δύναμη που αντιμετωπίζει το Άισι. Και είναι αλήθεια. Ήμουν και εγώ ήμουν και στο μέτωπο του Κυρκούρκ με τι ε, δυνάμει ε, των Κούρδων. Όμω οι δυνάμει. Ε, του Κουρδιστάν μεταξύ των οποίων αυτές του Μπατζάνι δεν κάνουν αυτή τη στιγμή εθνοκάθαρση με τους Γιαζίντι και τους Χριστιανούς ε, να απαλήφονται από περιοχές ολόκληρες αλλά και αραβικές ομάδες και ίσως όταν τελειώσουμε με, τον, με το Ισλαμικό κράτος, με το ISIS να βρούμε μπροστά μας μια πολύ σημαντική αντιπαράθεση μεταξύ Κούρδων, Αράβων, Τουρκμένων και Ασσύριων διότι οι άνθρωποι αυτοί θα έχουν ε, εκδιωχθεί από τι περιοχέ του με το πρόσχημα τη αντιμετώπιση του Άισι. Κάτι που είπε ένα συνάδελφο τώρα για το Ιρακινό στρατό. Ο Ιρακινό στρατό η Προσοντάμ Χουσέιν ήταν από του πιο δομημένου στρατού, από του πιο ικανού του αραβικού κόσμου και ίσω και από του καλύτερου του κόσμου. Γενικότερα, αυτή τη στιγμή ο στρατό δεν είναι ότι δεν είναι και τόσο επιχειρησιακό, είναι ότι δεν είναι καθόλου επιχειρησιακό ήμουν με τις μονάδες τις ευρωπαϊκές που, που έκαναν την εκπαίδευση των ειδικών δυνάμεων, εκπαίδευση των ειδικών δυνάμεων των Ιρακινών. Έτσι, τη μονάδα Σάικα και μου έλεγαν, στην πόλη του Σάικα μάλλον, και μου έλεγαν ότι ήταν πολύ κακή η επιχειρησιακή ε, δυνατότητα, η επικοινωνία ήταν πολύ κακή και ίσως να είναι μηδενική η επιχειρησιακή δυνατότητα τελικά. Υπάρχουν δύο μεγάλες νίκες στο Ραμάντι και στη Βαλούτζα. Στο Ραμάντι και στη Φαλούτζα όμως είχαμε μια αναλογία 6 προς 1 ή 10 προς 1. Και παρόλα αυτά αργήσαμε μήνες για να εκδιώξουμε το ISIS και με πολύ σημαντική ε, αεροπορική υποστήριξη. Ελικόπτερα επιθετικά που δεν άφηναν τις δυνάμεις του ISIS να κινηθούν. Όταν λοιπόν βλέπω αυτή τη νίκη όπου έχουμε μια αναλογία 6 προς 1, 10 προς 1 επαναλαμβάνω και με απόλυτη κυριαρχία στους αέρ, στον, στον αέρα ε, στους εθέρες επί μήνες, νομίζω ότι αυτό μας δίνει λόγους για να, να είμαστε αξιόπιστοι ως επιχειρησιακή δύναμη. Oh, okay, it seems, uh, the end... Πολύ ωραία. Δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις. ζητώ συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να κάνω μία ακόμα παρατήρηση μετά τα όσα είπε ο κύριος Φρόιντ. Σε καμία περίπτωση δεν θέτω να αμφιβόλω τα όσα είπατε, απλώς θα ήθελα να υπενθυμίσω κι εγώ μία εμπειρία που είχα. από τη δεκαετία του 90, στις αρχές μάλιστα της δεκαετίας του 90, στα πλαίσια της ε, Σολινταρνόσκα. Ήδη 35 χρόνια είχα περάσει εκεί. Μετά τις αλλαγές λοιπόν που είχαμε, τις πολιτικές στην ε, Πολωνία και μετά την νίκη της Πολυνταρνόσκα, μου δόθηκε η δυνατότητα να έρθω στις Βρυξέλλες και να συναντήσω άλλους συνδικαλιστές συναδέλφους εδώ στις Βρυξέλλες. και μολονότι νόμιζα τότε ότι είχα διεθνοποιηθεί, αν το θέσω έτσι, οτιδήποτε και αν σημαίνει αυτό, μου έκανε εντύπωση μία παρατήρηση που έκανε ένας συνάδελφος από το Τσάντ, που ήταν, είχε καταγωγή από το Τσάντ, ένας Αφρικανός συνάδελφος ο οποίος μιλούσε τότε για τον Σαντάμ Χουσέιν, που βέβαια βρισκόταν στην εξουσία τότε, και μου είπε, ξέρεις κάτι, είναι χειρότερος από το Χίτλερ, χειρότερος από το Χίτλερ. Και εγώ του είπα, ξέρεις τι σημαίνει αυτό το πράγμα για έναν Πολωνό, ξέρεις τι σημαίνει να λες έναν Πολωνό ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να είναι χειρότερος από το Χίτλερ. Πραγματικά σοκαρίστηκα, μπορώ να πω. Και η πρώτη μου αντίδραση ήταν «Μα πώς τολμάς να λες κάτι τέτοιο». Νομίζω ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είχε αρκετές γνώσεις τελικά, αλλά θυμάμαι ακόμα τα λόγια του αυτά. Μου εντυπώθηκαν ανεξίτηλα και αυτό το είπε ένας πολύ απλός άνθρωπος βασικά. Ένας άνθρωπος ο οποίος προερχόταν από τη Μαύρη Αφρική. Λοιπόν, Έχετε το λόγο. Ας δώσουμε πρώτα το λόγο στην κυρία Τζίλη και στη συνέχεια στον κύριο Κάουα Χασάν. Ευχαριστώ πολύ για όλες αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και παρατηρήσεις. Θα προσπαθήσω, προσπαθήσω να σας απαντήσω σε κάθε ερώτηση ξεχωριστά, ελπίζω. Ας ξεκινήσουμε από τις δικές σας ερωτήσεις, κυρία Πρόεδρε. Όσον αφορά τη φύση του Ισλαμικού κράτους, συμφωνώ με τον Καουά Χασάν, ο οποίος είπε ότι αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή μια παγκόσμια πρόκληση. Το ΝΤΑΕΣ δημιουργήθηκε στο Ιράκ, πήγε έπειτα στην Συρία και επικέντρωσε τη δράση του εκεί και πέστρεψε στη συνέχεια στο Ιράκ όταν του το επέτρεψαν βασικά οι περιστάσεις, όταν γίνανε πιο ευνοϊκές και θα έλεγα ότι όντω μοιάζει πλέον με ένα εμπορικό σήμα. Λειτουργεί σαν μάρκα, αν θέλετε. Και επομένω, όπω οποιοδήποτε μάρκα, είναι ευπροσάρμοστη, ευέλικτη. Και αυτή θα έλεγα ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Το ιδεολογικό ζήτημα, η ιδεολογική συνιστόσα είναι η πιο σημαντική και πιο κρίσιμη. και το γνωρίζουν αυτό. Ακολούθησαν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση επειδή αυτό τους ευνοούσε περισσότερο, επειδή σημείωναν κατά αυτόν τον τρόπο περισσότερες επιτυχίες και κέρδιζαν περισσότερο χρο... Ε, περισσότερη υποστήριξη. Θυμάστε ότι στην παρέμβασή μου στην αρχή είπα ότι θα μπορούσαμε τουλάχιστον πρόθεσμα να είμαστε αισιόδοξοι για την καταπολέμηση του Ισλαμικού κράτους, αλλά ότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε μπροστά μας ακόμα κάποιες μακροπρόθεσμες προκλήσεις, πολύ πιο σημαντικές ενδεχομένως και από το ίδιο το Ισλαμικό κράτος. Όντως μεταλλάσσεται το Ισλαμικό κράτος, έχει αυτή τη δυνατότητα, έχουμε ήδη δει αυτό, Προσπαθούμε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης να μην κάνουμε, αν θέλετε, τέτοιες προβλέψεις, αλλά ουσιαστικά αν το Ισλαμικό κράτος μπορεί κατά αυτόν τον τρόπο να κάνει επιθέσεις, επιθέσεις στη Βαγδάτη και με μία επίθεση να δολοφονεί 230 άτομα, αυτό σημαίνει βασικά ότι έχει αρχίσει πάλι να μεταλλάσσεται, ότι αλλάζει την τακτική του και ότι προχωρά αυτή τη στιγμή σε πιο παραδοσιακές μορφές πολέμου και επιθέσεων, ότι επικεντρώνεται εκ νέου σε στοχευμένες επιθέσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, και συμφωνώ εδώ πέρα με τον Καουά Χασάν, ότι θα πρέπει να δούμε το σφαιρικότερο πλαίσιο, το γενικότερο πλαίσιο, και όχι μόνο το Ιράκ και τη Συρία, αλλά όλη την περιοχή. Και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα φαινόμενο το οποίο αμφίβολα είναι παγκόσμιο, άρα και η πρόκληση είναι παγκοσμίων διαστάσεων. Θα προσπαθήσω να ομαδοποιήσω τώρα κάποιες ερωτήσεις. Αναφερθήκατε στο Βόρειο Ιράκ μας ρωτήσατε αν όντως ακολουθείτε μια πολιτική χωρίς αποκλεισμούς. Μας ρωτήσατε επίσης αν ήταν ενδεχομένω καλύτερη κατάσταση στο Ιράκ επί κυβέρνησης Σαντάμ Χουσέιν ή αν θα μπορούσαμε στο άμεσο μέλλον να δούμε μια χώρα που να λειτουργεί στην πράξη. Από τη θέση που έχω στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης Πιστεύω πραγματικά ότι η χώρα αυτή μπορεί να έχει μέλλον. Διαφορετικά θα άλλαζα θέση. Θα μπορούσαμε να δούμε τα πράγματα αισιόδοξα ή απεσιόδοξα, αλλά σε κάθε περίπτωση πιστεύω, είμαι πεπισμένη, ότι είναι δυνατό να καταλήξουμε σε μια καλώς λειτουργούσα χώρα, αλλά η πρόκληση είναι τεράστια. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο πιστεύω και εδώ συμφωνώ πάλι με τον συνάδελφό μου, είναι ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε σε κάθε περίπτωση με τις αρχές του Ιράκ. Το Ιράκ δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα μόνο του. Υπάρχει το ζήτημα των δυνατοτήτων, των ικανοτήτων, των θετικών επιρροών από άλλες χώρες, της υποστήριξης της διεθνούς κοινότητος. Και ακριβώς για όλα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να συνεχίσουμε να ζητάμε από όλους τους σημαντικούς παράγοντες της περιοχής να είναι παρόντες, να συμβάλλουν θετικά, να ασχολούνται με το Ιράκ και να μην αφιερώνε προσπάθειες στο Ιράκ μόνο κάθε φορά που γίνεται μια κάποια επίθεση. Όταν μιλάμε για συμφιλίωση, όταν μιλάμε για πολιτικές συμπερίληψεις, εστιαζόμαστε βασικά σε τομείς όπου θεωρούμε ότι χρειάζονται δύο παράλληλοι άξονες. Ένας άξονας ο οποίος ε, ξεκινάει από, τα, από τη βάση προς τα άνω, που θέλουμε να εμπλέξουμε βέβαια περισσότερο την κοινωνία των πολιτών. Θέλουμε δράσεις σε επίπεδο τοπικού πληθυσμού. Από το 2014 συγκεκριμένα και μετά βλέπουμε ότι υπάρχει μία πόλωση στην ε, Ιρακινή κοινωνία. Έχουν συμβεί διάφορα απέσια πράγματα, αποτρόπες εξελίξεις που δυστυχώς έχουν περάσει αρνητικά την κατάσταση και που ουσιαστικά μπορεί να οδηγήσουν σε εκδικητικές στάσεις από τις δύο πλευρές. Αυτό έχουμε δει και στη Φαλούτζα. Και αυτό είναι που μας ανησυχεί περισσότερο κάθε φορά που προσπαθούμε να δούμε τι θα απογίνει με τη Μοσούλη. Θέλουμε λοιπόν να προφήσουμε μια τέτοια στρατηγική bottom-up από τη βάση προς τα πάνω, εμπλέκοντας την κοινωνία των πολιτών, αλλά θα καταφέρουμε να πετύχουμε, αν θέλετε, την στρατηγική μας αυτή, αν υπάρχει και η αντίστροφη τάση από τάνω προς τα κάτω δηλαδή. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο σε όλα τα συμπεράσματα, για παράδειγμα του Συμβουλίου, σε όλες τις δηλώσεις που κάνουμε, λέμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, όλοι οι πολιτικοί και οι θρησκευτικοί ηγέτες να αρχίσουν να συνεργάζονται με απότερο σκοπό τη συμφιλίωση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα του στρατού. Ναι, όντως, το ζήτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό. και νομίζω ότι νομιμοποιήστε απόλυτα να θέτετε το ερώτημα αυτό και όλοι αυτό ουσιαστικά ρωτούν από το 2014 και μετά όταν είδαμε ότι άρχισε να αποσύρεται τελικά ο στρατός, να εγκαταλείπει τα όπλα του στη Μοσούλη. Ποια είναι τώρα η δική μας άποψη. Θεωρούμε ότι αυτό συνδέεται κυρίως με την πολιτική κατάσταση της χώρας. Έτσι εξηγούνται τα φαινόμενα αυτά. στο Ιράκ. Δεν υφίσταται πλέον ένας ισχυρός εθνικισμός ή ένας ε, ισχυρός εθνικός ιστός, αν θέλετε, με τη θετική έννοια του όρου. Δεν υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει συνεκτικότητα ανάμεσα στον πληθυσμό. Ορισμένοι θα πούν ότι το ζήτημα δεν είναι καν η κατάρτιση, αλλά η ίδια η πολιτική βούληση, η βούληση αν θέλετε, και πολλές φορές ακόμα και στα πλαίσια του στρατού δεν υπήρχε η απαραίτητη βούληση, κυρίως ε, από τους ε, ΣΥΙΤΕΣ, να πεθάνουν αν θέλετε για τη Μοσούλη, να δώσουν τη ζωή τους για μια τέτοια μάχη. Υπάρχουν ορισμένοι που λένε ότι οι δυνάμεις λαϊκής κινητοποίησης, αυτές οι λαϊκές πολιτοφυλακές PMF, λειτουργούν καλύτερα, ότι είναι πιο αποτελεσματικές. Στην πράξη όμως, και αυτό που έχουμε δει πρόσφατα, είναι ότι οι ομάδες PMF τελικά μάλλον είναι και πιο κινητοποιημένες. Έχουν πιο ισχυρή βούληση. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο χρειαζόμαστε περισσότερο κράτος, πιο ισχυρές κρατικές δομές, προκειμένου να καταφέρουμε να αποκαταστήσουμε, αν θέλετε, ένα κοινωνικό σύμφωνο με τον πληθυσμό. Και μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα θετικό εθνικό πνεύμα στη χώρα. Τώρα, η κατάσταση του Κορδιστάν και γενικότερα το βόρειο τμήμα της χώρας. Αναφέρθηκα ήδη σε αυτό. Σας είπα ποια είναι η απόψή μας. Πού βασίζεται τώρα αυτή η απόψή μας. Επί του παρόντος δεν νομίζουμε ότι οποιαδήποτε κοινότητα στο Ιράκα είναι σε θέση να διαχειριστεί το κράτος ή κάποιο τμήμα του κράτους. Συνεπώς, Επί του παρόντος, η μόνη λύση είναι να έχουμε πραγματικά ένα συνασπισμό και όλοι μαζί να καταφέρουμε να οικοδομήσουμε αυτή τη χώρα. Τα ό,τι συνέβησαν στην Μοσούλη ουσιαστικά εξηγούνται από το ότι στο βόρειο τμήμα της χώρας από το 2003 και μετά, ενδεχομένως και πριν από το 2003, δεν υπήρχε συγκεκριμένος έλεγχος από την κεντρική κυβέρνηση. Ήταν μια ζώνη εκτός ελέγχου, αν θέλετε. Το ίδιο ισχύει και για την Άμπα, όπου ουσιαστικά είχαμε θύλακες μέσα στη χώρα που ξέφευγαν από κάθε πιθανό κρατικό έλεγχο. Κατά την άποψή μας, λοιπόν, αυτό το οποίο θα μπορούσε να επιφέρει μια πιο βιώσιμη λύση είναι να επαναφέρουμε το κράτος στις περιοχές αυτές αντί να λέμε ότι ο διαχωρισμός της χώρας σε επιμέρους τμήματα θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Η διάσπαση της χώρας αυτή τη στιγμή, ιδίως δεδομένη της υφιστάμενης κατάστασης, θα είχε πολύ αρνητικές επιπτώσεις. Ο κατακαιρματισμός ήδη υπάρχει σε επίπεδο πολιτικό, αλλά και σε επίπεδο κοινωνία στη χώρα. Η διάσπαση λοιπόν περαιτέρω της χώρας θα έχει πολύ αρνητικές δευτερογενείς συνέπειες. Τώρα, η επιρροή άλλων σημαντικών παραγόντων της περιοχής. Σαφώς υπάρχει τέτοια επιρροή. Θυμάμαι ότι ορισμένοι συνάδελφοι είχαν πει στο παρελθόν ότι το Ιράν είναι πανταχού παρόν στο Ιράκ. και ότι είχαν ε, αναλάβει κατά κάποιο τρόπο την διαχείριση διαφόρων εκστρατιών στο Ιράκ. Αν υπάρχει πράγματι μία χώρα που ενδιαφέρεται τόσο και εμείς για το Ιράκ είναι το Ιράν. Αν υπάρχει μια χώρα που όλοι οι σημαντικοί διεθνείς παράγοντες εμπλέκονται και έχουν κοινά συμφέροντα, αυτό είναι το Ιράκ. Ο κατακαιρματισμός, η αστάθεια, ο διαχωρισμός της χώρας προφανώς δεν συμφέρει κανέναν απολύτως. Δεν είναι προ το συμφέρον του Ιράν, δεν είναι προ συμφέρον τη Σαουδική Αραβία, δεν λειτουργεί προ το συμφέρον τη Τουρκία, καμία τελικά χώρα. Επομένω, ενδεχομένω θα πρέπει να επικεντρωθούμε εκεί που έχουμε όντω ένα κοινό συμφέρον, δηλαδή στο Ιράκ, και να προσπαθήσουμε να δούμε πώ μπορούμε να πειράσουμε θετικώ τα πράγματα, χωρί όμω να είμαστε αφελεί. Γιατί βέβαια γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή σε εξασφαλίσει κανεί μια κάποια επιρροή, είναι πολύ δύσκολο να σταματήσει μετά ή να παραμείνει ουδέτερο. Ακριβώ όμω επειδή υπάρχουν τόσα πολλά διαφορετικά συμφέροντα και ουσιαστικά ένα κοινό συμφέρον υπέρ του Ιράκ, αν καταφέρουμε όλοι από κοινού να διατηρήσουμε την ενότητα της χώρας, τότε θα καταφέρουμε να βρούμε και μια ισορροπημένη λύση όσον αφορά τις αρμοδιότητες που θα μπορούσαν να λάβουν οι περιφερειακοί παράγοντες. Νομίζω ότι κάλυψα τις περισσότερες ερωτήσεις ο κύριος Χασάν. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για όλες αυτές τις ερωτήσεις, για όλες αυτές τις παρατηρήσεις. Ήταν όντως πολύ εύστοχες ερωτήσεις. Δυστυχώς δεν έχω απαντήσεις για όλες. Όπως είπε και η Ρόζα Μαρία, ενδεχομένως να δημιουργούμε περισσότερες ερωτήσεις παρά να μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα επί του παρόντος με το Ιράκ. Να ξεκινήσω με το ζήτημα της αλληλεγγύης, κυρία Πρόεδρε. Όντως, είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή υπήρχαν σημαντικά μηνύματα αλληλεγγύης υπέρ του Ιράκ από πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Θα έλεγα όμως ότι το πιο σημαντικό να μιλήσουμε για την κοινωνική πτυχή της αλληλεγγύης. Αλληλεγγύη προς την κοινωνία. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ενώσουμε, αν θέλετε, τι διαφορετικέ κοινωνίε μεταξύ του. Για ποιο λόγο να μην τηρήσουμε ενό λεπτού στη γη και τα θύματα τη Δάκα ή τη Καράντα ή τη Κωνσταντινούπολη. Θα μπορούσαν, ε, για παράδειγμα, οργανισμοί ε, στο Βέλγιο ή σε άλλες χώρες να λάβουν μια τέτοια πρωτοβουλία. Αυτό πραγματικά θα αποτελούσε μια πολύ σημαντική συμβολική υποστήριξη προς τα θύματα που έχουμε στο Ιράκ, ε, συγκεκριμένα στη Βαγδάτη και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Αυτό είναι εξίσου σημαντικό και εξίσου ισχυρό με οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση. Θετικά νέα και θετικές εξελίξεις, ναι, προφανώς υπάρχουν. Έχουμε κυρίως αρνητικές ειδήσει από το Ιράκ, αλλά εγώ προσπαθώ μελετώντας τη χώρα αυτή να βλέπω και τις δύο πλευρές. Θετικές εξελίξεις μπορούμε να έχουμε στο Κουρδιστάν και σε άλλες περιοχές του Ιράκ που επισκιάζονται όμως από τις καθημερινές εκφάνσεις βαρβαρότητας του Ισλαμικού κράτους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταπολεμά κανείς σε καθημερινή βάση ένα τεράστιο εχθρό όπως το ISIS. Αυτό επισκιάζει από μόνο του οποιαδήποτε θετική εξέλιξη θα μπορούσαμε να είχαμε στη χώρα. Θα σα δώσω κάποια θετικά παραδείγματα. Για παράδειγμα, είχαμε διαδηλώσει στην Παγδάτη πριν από δύο μήνες που παρουσιάστηκαν από κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης της περιοχής αλλά και διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μονομερός όμως αυτό δεν ίσχυε. Δεν ίσχυε κάτι τέτοιο υπήρχαν άνθρωποι από, όχι μόνο από το Σάντερ, αλλά και από άλλες τάσεις και άνθρωποι οι οποίοι δεν ανήκαν σε κάποιο πολιτικό κόμμα και που απλώς θέλανε να προωθήσουν περισσότερο μια πιο ενωπημένη ιδέα της κοινωνίας και του κράτους. Άνθρωποι οι οποίοι δεν ανήκαν αγκαστικά σε κάποια πολιτικά κόμματα ή κινήματα. Και άνθρωποι αυτοί κατέβηκαν στους δρόμους της Βαγδάτης και ζητούσαν περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη λογοδοσία Θέλαν να γνωρίσουν ακριβώς τι συνέβη με την επίθεση στην Καράντα, ποιος ήταν ο υπεύθυνο. Δυστυχώς όμως το μήνυμα αυτό δεν πέρασε στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης και δεν έφτασε και σε εμά βέβαια, έτσι δεν είναι. Έχουμε λοιπόν όντω έναν έντονο ακτιβισμό στο Κουρδιστάν, στην Πασρά, από την κοινωνία των πολιτών, άνθρωποι οι οποίοι ζητάνε πραγματικέ μεταρρυθμίσει, χρηστή διακυβέρνηση, απευθύνεται στις κουρδικές και ιρακινές αρχές να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες. Δυστυχώς όμως δεν το μαθαίνουμε αυτό, ακριβώς επειδή επισκιάζεται από το συνεχή πόλεμο κατά του Ισλαμικού κράτους. Όσον αφορά τώρα το στρατό και θα το συνδέσω αυτό και με την έκθεση Τζιλ Κόρπτες στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι σε καλύτερη κατάσταση το Ιράκ σήμερα από ό,τι στο παρελθόν μετά το 2003. Η έκθεση δεν ε, κοινοποιήθηκε στο Ιράκ. Δεν, μάλλον δεν συζητήθηκε καν στη χώρα αυτή. Ε, ακούστηκε κάπως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά τίποτα παραπάνω. Νομίζω ότι οι ίδιοι Ιρακινοί έχουν ξεπεράσει, αν θέλετε, την εποχή εκείνη. Και ας μην ξεχνάμε ότι σε καμία περίπτωση η σταθερότητα η οποία προέρχεται από ένα αυταρχικό κράτος δεν είναι πραγματική σταθερότητα. Το έχουμε δει αυτό σε πάρα πολλές περιοχές. Στην Τινησία, στη Λιβύη, στη Γεμένη. Πάντα η επισφαλής αυτή σταθερότητα τελικά οδηγεί σε εξεγέρσεις. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να επηρεαζόμαστε αυτή τη στιγμή από τα όσα βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Υπήρχε κρατική τρομοκρατία την εποχή του Σαντάμ Χουσέιν. Αυτή τη στιγμή η τρομοκρατία, αν θέλετε, είναι πολυσχηδής και τελικά επισκιάζεται πάρα πολύ από τις ε, βαρβαρότητες του Ισλαμικού κράτους. Καταλαβαίνω λοιπόν αυτούς οι οποίοι υποστηρίζουν την άποψη την οποία εκθέσατε και μάλιστα υπήρχε και ένα ρεπορτάζ στο αραβικό BBC, μια συνέντευξη με τον άνθρωπο αυτό που το 2003 είχε ρίξει το άγαλμα του Σαντάμ Χουσέιν, που το είδαμε όλοι στι ειδήσει, και ουσιαστικά έλεγε αυτή τη στιγμή ότι μετανιώνει για την πράξη του εκείνη, για τι εξελίξει εκείνη τη εποχή, γιατί βλέπει ότι επί του παρόντο στη χώρα του δεν υπάρχει σταθερότητα. Αν όμω ο Σαντάμ Χουσέιν ήταν ακόμα στην εξουσία, τι είδου Ιράκ θα είχαμε σήμερα. Νομίζω θα βλέπουμε περισσότερα φαινόμενα γενοκτονία, χρησιμοποίηση χημικών όπλων κατά διαφόρων ομάδων και κοινοτήτων, και η οικογένεια του Σαντάμ Χουσέιν, η γη του, οι κόρε του, θα βρισκόταν στην εξουσία, στην για τα επόμενα 50 χρόνια. Επομένω, α μην θεωρούμε ότι η περίοδο πριν από το 2003 ήταν εφετική. Όσον αφορά τώρα τους Κούρδους, το βόρειο τμήμα της χώρας, νομίζω ότι υπάρχει μια παρανόηση εδώ. Δεν είπα ότι οι Κούρδοι προχώρησαν σε εκάθαρση. Αυτό που είπα είναι ότι στη Σιντζάρ οι Γεζίντις, είναι θύματα της ε, διαμάχης που έχουμε ανάμεσα σε KDP και PKK. Αυτό είναι πραγματικότητα όμως. Ξέρετε ότι υπάρχουν πολιορκίες και οικονομικά μπλόκα, ακριβώς επειδή αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εσωτερική διαμάχη ανάμεσα σε KDP και PKK. Δεν περίμεναν οι Γεζίδοι να δούνε κάτι τέτοιο επιστρέφοντας όμως στην ιδιαίτερη πατρίδα τους τη στιγμή που έφυγε το ISIS. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει ε, κατανομή των εξουσιών, των αρμοδιοτήτων και μεταξύ της περιοχής αυτής και μεταξύ της Βαγδάτης. Οι κουρδικές δυνάμεις θα πρέπει να καταλήξουν σε ένα κοινό όραμα, να επιλύσουν τις μεταξύ τους διαφορές και να έχουν πλέον ένα συγκεκριμένο σχέδιο για να δούνε πώς θα εξελιχθεί τελικά και το Ιράκ αλλά και η περιοχή του Κουρδιστάν. Για το αν είναι δυνατόν ένα άλλο Ιράκ. Να πω πρώτα απ' όλα το εξή. Η εναλλακτική σε ένα ειρηνικό Ιράκ και θα με όμως είναι δεκαετίες εμφυλίων πολέμων μεταξύ και εντός των κοινοτήτων ότι ήταν ο Λίβανος ε, τη δεκαετία του 70 και του 80 δεν θα είναι τίποτα σε σύγκριση με το Ιράκ. Αυτή είναι η εναλλακτική. Και δεν θέλω να κινδυνολογώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η πολιτικοστρατιωτική πραγματικότητα. Δεν υπάρχει εναλλακτική από το να ε, εμπλακούν οι Ιρακινοί. Αυτοί πρέπει να κάνουν δύσκολη δουλειά, αλλά χρειάζονται τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μακροχρόνια εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της διεθνούς κοινότητας, να πιέσει τους Ιρακινούς να συνεννοηθούν και να καταλήξουν σε κάποια συνένεση. Τι οι Ιράκ θέλουν. Κατά την άποψή μου δεν θα επανέλθουμε στην κατάσταση του πολιτικού συστήματος πρώτου 2003. Αυτό το οποίο θα προκύψει και πάλι με βάση τα όσα συμβαίνουν επί είναι ε, μια ομοσπονδία ή και συνομοσπονδία ακόμα. Είναι δύσκολο αυτό. Χρειάζεται πολλές διαπραγματεύσεις, αλλά και διεθνή εμπλοκή και μεσολάβηση, γιατί δεν μπορούν να το κάνουν μόνοι τους οι Ιρακινοί. Και δεν είναι μόνο ζήτημα του Ιράκ, είναι διεθνές. Είναι λοιπόν προς το μακροπρόθεσμο συμφέρον της Ένωσης ε, να παραμείνει ε, εκεί και να μεσολαβήσει μεταξύ Κούρδων, μεταξύ Κούρδων και Αράβων, μεταξύ Σουνιτών, Σιητών και λοιπόν και θα χρειαστεί ε, χρόνο, δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να γίνει. Και μιλώντας για το εάν είναι δυνατό, δυνατό ένα άλλο Ιράκ. Οι Ιρακινοί πρέπει να συμφωνήσουν για ένα μεταβατικό σχέδιο για τα επόμενα 5-10 χρόνια για να αναπτυχθούν τα πλαίσια ενός νέου κράτους, είτε ομοσπονδιακού είτε συνομοσπονδιακού και θα πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το μοντέλο. Αλλά δεν μπορούμε να αποφύγουμε την ε, ανάγκη ενός μεταβατικού σχεδίου τουλάχιστον για 5-10 χρόνια και να δούμε πώς οι κοινότητες και τα κόμματα του Ιράκ θα αντιμετωπίσουν αυτό το νέο κράτος, ποιοι δεν θέλουν να λειτουργήσει, ποιοι είναι οι πραγματικοί ηγέτες που νοιάζονται για το Ιράκ και τις διάφορες επαρχίες και μόνο έτσι μπορούμε να κρίνουμε το πώς θα πάει η διαδικασία. Αυτά. Θα επανέλθω μετά σε άλλα ζητήματα. Κοιτάξτε, νομίζω πως υπάρχουν ίσως ερωτήσεις. Ε, ναι, κύριε Φρόιντ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να ξεκαθαρίσω το εξής για να μην παρεξηγούμε. Με το να μεταφέρω τα λόγια του Τόνι Μπλερ δεν ήθελα οπωσδήποτε να υπονοήσω ότι ε, νοσταλγώ τα όσα συνέβησαν επί Σαντάμ Χουσέιν γιατί κάνατε αυτή την ε, παρομοίωση με το Τσάντ δεν ξέρω από πού προέκυψε αυτό δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου. Ελπίζω να μην παρεξηγήθηκα. Θα ήθελα να κάνω κι εγώ άλλη μια ερώτηση πολύ συγκεκριμένη και οφείλεται στο ιδιαίτερό μου ενδιαφέρον. Θεωρείτε και οι δυο σας ότι με αυτό το πενταετές μεταβατικό σχέδιο υπάρχει περιθώριο για την επιστροφή των ε, χριστιανών. Υπήρχαν τρομερές ακρότητες και εγώ επειδή γνωρίζω αρκετούς από αυτούς. Η Μέση Ανατολή ήταν το λίκνο οπωσδήποτε του χριστιανισμού ε, τώρα είναι πια μειονότητα και ε, τόσο για πολλά χρόνια ήταν ειρηνική η κατάσταση. Ναι, εντάξει. Υπήρχαν βεβαίως ε, κάποια σκαμπανεβάσματα, αλλά σε σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν ήταν μια ειρηνική συνύπαρξη. Θεωρείτε ότι στο προσεχές μέλλον θα υπάρχει χώρος για αυτές τις εξελίξεις ή ήταν επιτυχής αυτή η εθνική εκαθάριση. Σας ευχαριστώ. Η επιστροφή χριστιανών και λοιπόν, γεζίτιδων και λοιπόν. Ξέρετε όταν μιλάω με τους φίλους μου γεζίτιδες χριστιανούς και λοιπούς που έφυγαν είναι ακόμα στο Ιράκ. Ήμουν πριν από λίγου μήνε στο Κουρδιστάν και συνάντησα εκεί κάποιου ε, γεζίτιδε. Κάποιοι θέλουν να φύγουν τελείω, Δεν θέλουν να επιστρέψουν, έχουν περάσει όσα πέρασαν. Άλλοι θέλουν να επιστρέψουν ε, υπό την προπόθεση ότι θα υπάρχει κάποια χρηστή διοίκηση. Θα μπορούν και αυτοί να έχουν λόγο στο ποιο ε, κυβερνά την περιοχή τους. Και αυτά δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Πρέπει λοιπόν να επιμείνουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στις ε, τοπικές αρχές, ε, στην Ιρακινή κυβέρνηση, στις κουρδικές αρχές, πως όσον αφορά τους εσωτερικά εκτοπισμένους, πρέπει να υπάρξουν κάποιες εγγυήσει ότι θα υπάρξει αυτοδιοίκηση σε περιφερειακό επίπεδο, θα υπάρξει χρηστή διοίκηση και όσον αφορά την εσωτερική ασφάλεια θα μπορούσαν δικοί τους άνθρωποι να εγγυώνται την ε, ασφάλεια. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι φοβάμαι ότι περισσότεροι από αυτούς δεν θα επανέλθουν, δεν θα επιστρέψουν μόνιμα. Ε, για το θέμα του στρατού και των υπηρεσιών ασφαλείας. Ξέχασα να το πω. Ναι, πραγματικά κατέρευσε ο στρατός ε, του 2014. Ε, είναι γεγονός αυτό, αλλά ταυτόχρονα ο στρατός πριν από μια εβδομάδα κατέλαβε μια πόλη με την υποστήριξη οπωσδήποτε της Αμερικανικής αεροπορίας. Ε, αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική. Πρέπει να υποστηριχθούν οι Πεσμεργά, οι PMS για να, να καταλάβουν τις πόλεις. Ο λεγόμενος νόμος περί εθνοφρουράς που μπλοκάρεται στο κοινοβούλιο του Ιράκ και ίσως πρέπει να σας απασχολήσει στη συζήτηση σας ε, με τις αρχές. Προβλέπει οι ε, διοικητές των περιφερειών ε, να έχουν τις δικές τους εθνοφρουρές σε κάθε περιφέρεια και επίσης να, δημιουργηθεί, να δημιουργηθούν περιφερειακές αστυνομίες και υπηρεσίες ασφαλείας για τα θέματα αυτά. Οπότε έτσι θα καλυφθεί το ζήτημα αυτό της επιστροφής του στρατού στις διάφορες επαρχίες. Ξέρω πως ο κύριος Νάρτη ήθελε τον λόγο. Ναι, συντομία. Εγώ έχω σχέση με μέλη των, της κοινότητας των Συρίων, ε, των Γιαζίντι, της κοινότητας των Σουνιτών στο Βόρειο Ιράκ και η πραγματικότητα είναι ότι βεβαίως όταν υπάρχει σύραξη, όταν υπάρχει πόλεμος κάπου, ο κόσμος φεύγει. Και όταν τελειώνει ο πόλεμος, επιστρέφουν όσοι μπορούν και όπου μπορούν. Η πραγματικότητα όμως επίσης είναι και μου τη διηγήθηκαν και θα πάω και επί τόπου και θα τη διαπιστώσω και αυτό το άκουσα ομόφωνα από όλους είναι ότι με αφορμή τον πόλεμο σε περιοχές όπου θα μπορούσαν κάλλιστα να επιστρέψουν, δεν μπορούν να επιστρέψουν. Και υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες, έτσι ώστε οι υπόλοιπε κοινότητες που βρίσκονται στα όρη Σιντζάρ να μπορέσουν να επιστρέψουν. Διότι σε μια τόσο στρατηγική περιοχή όπως την περιοχή του Σιντζάρ, δηλαδή είναι όλος ο βόρειος διάδρομος για το Κουρδιστάν, είναι σημαντικό να παραμείνει αυτός ο διάδρομος. Αν δει κανείς το χάρτη της Συρίας, παραδείγματος χάρη, καταλαβαίνει ότι η κουρδική κοινότητα βρισκόταν μόνο στην Δύση. Υπήρχε μόνο και το Άριαν Άραπ, το Κομπάνε και το Ισκεντερούμ κοντά στην Αλεξανδρέτα. Δηλαδή, τώρα υπάρχει ε, ένα σημα... ένας συνεχόμενος διάδρομος και αυτό από στρατηγική πλευρά είναι σημαντικό. Εάν δείτε επίση ότι όλε οι δηλώσει που κάνουν οι Κούρδοι ηγέτε είναι ότι απελευθέρωση, τα απελευθερωμένα εδάφη από, πεσ, Πεσμεργά θεωρούνται κουρδικά εδάφη και ότι στο Κυρκούρκ υπάρχει κουρδικοποίηση και αποκλεισμό των αραβικών και των τουρκμενικών κοινοτήτων ε, μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει βούληση από πλευρά Κουρδιστάν ε, να γίνει κάτι άλλο από μια εθνοκάθαρση ή εν την, ε, την παρεμπόδια της επιστροφής που είναι το ίδιο όποιος δεν το βλέπει αυτό δεν είναι σε επαφή με την πραγματικότητα υπάρχει λοιπόν ηγεμονία από τους Κούρδους de facto έχουν αρχίσει να προσαρτούν περιοχές που δεν ήταν ποτέ κουρδικές ή που ήταν κουρδικές ιστορικά και που θέλουν πλέον να ανακτήσουν. Υπήρξαν περιοχές απικιοποίηση αραβικής ήταν και σχέδιο του να είναι αυτό το Κυρκούρκ αλλά σιγά σιγά αφήνουμε εκτός οποιοδήποτε κοινότητα μη κουρδική οπότε αυτό είτε το θέλουμε είτε όχι θα, θα οδηγήσει σε νέες, θα οδηγήσει σε νέες σειράξεις και σε έναν επόμενο πόλεμο well, I think it is worth... Νομίζω πως ε, αξίζει να τα σχολιάσετε. Λοιπόν, ε, δεν ξέρω ποιος ε, θέλει, είναι και οι δύο. Α, ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα κατάλαβα, γιατί παρεξήγησα όταν μιλήσετε για εθνικές εκαθαρίσεις, τώρα κατάλαβα. Γιατί δεν ήταν σαφές στην πρώτη σας παρέμβαση. Αν κάνουν εθνικές καθαρίσεις οι Κούρδοι. Σύμφωνα με κάποιες εκθέσεις της Human Rights Watch υπήρχαν κάποια ζητήματα σε κάποιες περιοχές και οι κουρδικές αρχές είπαν ότι λόγω της φύσης του πολέμου σε περιοχές αυτές ανεξαρτήτως του ποια είναι η αλήθεια νομίζω και το είπα ότι υπάρχει η ανάγκη πρώτα απ' όλα ε, όποιος και αν έκανε κάτι τέτοιο είναι έγκλημα δεν, δεν πρέπει να να συμβαίνει όποιος και αν το κάνει ε, Σιήτες, Σουνίτες, Κούρδοι. Και το αποτέλεσμα είναι ακόμη περισσότερη ριζοσπαστικοποίηση. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Όταν μιλάμε τώρα για αμφισβητούμενες περιοχές, Κυρκούκ, Μοσούλη και αλλού, και πάλι επανέρχομαι σε αυτό το οποίο είπα. Υπάρχει ανάγκη σοβαρών διαπραγματεύσεων μεταξύ της ε, περιφερειακής κυβέρνησης του Κουρδιστάν και της Βαγδάτης με εμπλοκή του ΟΗΕ, των ΙΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καταλήξουν σε έναν συμβιβασμό και να κάνουν ένα μεταβατικό σχέδιο για τα επόμενα 5-10 χρόνια. Μόνο έτσι θα λυθεί αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Εσείς, ναι. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσω. Ε, δεν είμαστε τυφλοί. Βεβαίως έχουμε πληροφορίες για τα όσα συμβαίνουν στη χώρα και χρησιμοποιούμε και η υπατή εκπρόσωπος ε, τον πιο διπλωματικό όρο δημογραφική μηχανική που είναι αυτό το οποίο συμβαίνει παντού στη χώρα. Και γι' αυτό επιμένουμε τόσο πολύ στον σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, του κράτους δικαίου, αντιλαμβανόμενοι ότι πρέπει να είναι μια επιλογή τοπική των ανθρώπων στη χώρα θεωρούμε ότι ένας μεταβατικός μηχανισμός δικαιοσύνης που θα είναι αποδεκτός από τους Ιρακινούς ε, στο μέλλον θα είναι κάτι το οποίο θα παίξει ρόλο κλειδί στην συμφιλίωση γιατί γνωρίζουμε ε, το τι συμβαίνει και είναι πράγματι φρικτό. Ε, δεν χρειάζεται να είμαστε αφελείς. Πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο κάνουμε, να στέλνουμε τα μηνύματα, να απευθύνουμε εκκλήσεις στους διάφορους ηγέτες να φανούν υπεύθυνοι. Τώρα, αν θα επιστρέψουν οι χριστιανοί και οι άλλες μειονότητες. Είναι πρόβλημα για τις μειονότητες, αλλά έχει γίνει και για την Παγδάτη ε, από ό,τι βλέπουμε. Με ρώτησαν ε, κάποτε τι θα έκανες ε, αν ήσουν ε, Ιρακινοί και ήσουν στη Βαγδάτη. Και είπα, «Ε, ε, προσπαθήστε να μείνετε, η χώρα σας, σας χρειάζεται. Και ήρθε ο ίδιος άνθρωπος μετά από έξι μήνες και μου είπε θέλω μια βίζα για... πήρα βίζα για τη Γερμανία και θα πάω στη Γερμανία και δεν θα ξαναγυρίσω ποτέ. Οπότε εξαρτάται από τις συνθήκες που επικρατούν και εξαρτάται από το αν υπάρχει ελπίδα. Αν υπάρχει ελπίδα, ε, ο κόσμος μπορεί να λέει ότι θα επιστρέψει, αλλά τη στιγμή που θα αντιληφθούν ότι η χώρα μπορεί να ξανακυλήσει σε έναν τρομερό εμφύλιο πόλεμο, και συμφωνώ εδώ πέρα μαζί σας ότι αν πάνε προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι πολύ χειρότεροι από ό,τι είχαμε δει στο Λίβανο και στα Βαλκάνια. Γιατί αυτό το οποίο διακυβεύεται και από πλευράς ε, συμφερόντων είναι τεράστιο στο Ιράκ. Εξαρτάται λοιπόν από την ικανότητα των Ιρακινών αρχών πρώτα απ' όλα και την στήριξη της διεθνούς κοινότητας να δώσει κάποια ελπίδα σε αυτούς τους ανθρώπους γιατί είναι σαφές ότι αν έχουν κάποια επιλογή θα μείνουν εκεί. Μια τελευταία λέξη για το αν το Ιράκ είναι καλύτερα πριν ή μετά τον Σαντάμ. Θα έλεγα πως μια χτίδα ελπίδας που φάνηκε είναι ότι παρόλα αυτά έχουν κάτι το οποίο δεν είχαν πριν είναι ότι έχουν μια εμβριακή δημοκρατία μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα μέσω δημοκρατικών διαδικασιών και αυτό μας κάνει να ελπίζουμε ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Και το εξής, ότι έχουν ε, ένα υψηλό επίπεδο για το τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί στη χώρα και σε σύγκριση και με τις ε, χώρες της ε, περιοχής. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήταν συναρπαστική η συζήτηση. Θα συνεχίσουμε μετά την επιστροφή μας από το Ιράκ γιατί γίνεται και μια συζήτηση μετά την αποστολή. Και το ενδιαφέρον μας ε, για την ευημερία του Ιράκ είναι συνεχές. παρά το ότι η διεθνή κοινότητα ε, όπως αστειευόμαστε ε, μπορεί να αντιμετωπίζει μόνο ένα δύσκολο ζήτημα τη φορά και υπάρχουν πολλά ε, δύσκολα ζητήματα που... αυτά το ενδιαφέρον μας για το Ιράκ είναι συνεχές και αδιακόπα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την πολύ συναρπαστική συζήτηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους βουλευτές που συμμετείχαν, το προσωπικό και τέλος βεβαίω τους διερμηνείς. Ήταν μια δύσκολη συνεδρίαση αλλά πολύ ενδιαφέρουσα. Σας ευχαριστώ. Τελειώσαμε με αυτό το σημείο. Το τελευταίο είναι τα διάφορα. Ελπίζω να μην υπάρχει τίποτα. Η επόμενη συνεδρίαση είναι στις 5 Σεπτεμβρίου. Καλές διακοπές. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.